κάτι το οποίο θα παραμείνει σημαντικό και όλοι νομίζω ότι έχουμε κοινού στόχους σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ λοιπόν. Κλείνουμε την συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει από τις 12 και μετά σε λίγα λεπτά. Το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι η έκθεση για το πώς θα αποφύγουμε τη, δαπάνη, τη σπατάλη των τροφίμων. Να σας πω ότι η συζήτηση αυτή ε, είναι πολύ σημαντική η τηλεόραση της ε, χώρας μου αφιέρωσε πάρα πολλές εκπομπές για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ήδη αγγίζει την ε, κοινή γνώμη, κάτι το οποίο σπάνια συμβαίνει σε σχέση με τις δικές μας συζητήσεις. Έχει το λόγο ο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της σύνταξης αυτής ε, της έκθεσης. Ήταν θα έλεγα μία όριμη προσπάθεια η οποία θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε στο θέμα το τι θα κάνουμε με, την, ε, με τα ε, τρόφιμα αυτά τα οποία δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα με σωστό τρόπο. Πράγματι είναι αλήθεια ότι, έχουν, ε, ε, ε, ότι είναι σαφές ότι ένα από τα κυριότερα προβλήματα του άμεσου μέλλοντος θα είναι να αντιμετωπιστεί μια μεγάλη και ιδιαίτερα σημαντική απέτηση για τρόφιμα. Και επομένως το θέμα της διατροφικής ασφάλειας έχει γίνει ένα από τα δυσκολότερα ως προς την αντιμετώπιση του. Και επομένως εμείς δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε σε αυτούς να παραμείνουμε αδρανείς απέναντι σε αυτό το φαινόμενο δηλαδή τη πατάλης των τροφίμων. Όταν αναφερόμαστε σε τρόφιμα, αναφερόμαστε σε τρόφιμα τα οποία είναι απολύτω βρόσιμα ακόμα, είναι σε απόλυτα άριστη κατάσταση στην ουσία έχουμε φτάσει πλέον σε ένα τέτοιο ε, επίπεδο που η ΦΑΟ θεωρεί και εκτιμά ότι ένα τρίτο των ε, τροφίμων ε, σπαταλιέται από τα τρόφιμα τα οποία προσφέρονται στην ανθρώπινη κατανάλωση. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα τέτοιο επίπεδο που πρέπει να πούμε ότι πλέον δεν αντιμετώπιζουμε μονάχα ένα ηθικό δεοντολογικό πρόβλημα αλλά ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα με μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν και με τούτη την ε, έκθεση προσπαθούμε να πείσουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να βάλει στην ημερήσια διάταξή της, στην πολιτική της ατζέντα, το ζήτημα της σπατάλης των τροφίμων θα πρέπει να εξευρεθεί κοινή στρατηγική έτσι ώστε να κάνουμε αυτήν, αυτό το άλμα ποιότητος το οποίο ε, θα ε, ε, μας οδηγήσει σε σημαντική μείωση της πατάλη των τροφίμων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε με όλα τα κέντρα πρωτοβουλειών, οργανώσεις, εθελοντές κλπ που έχουν απτά προγράμματα στο ζήτημα αυτό σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις που έχουν έχουν ε, εξοικονομηθεί ε, τρόφιμα τα οποία έχουν δοθεί ε, στους ευάλωτους πληθυσμούς της Ευρώπης. Είναι εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Γι' αυτό ζητούμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεκριμένα μέτρα. Κυρίως να τροποποιηθούν οι κανονισμοί για, τις, για τους δημόσιους διαγωνισμούς, για τη μαζική εστίαση, τις ε, ε, καντίνες κτλ. Να έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο ε, θα είναι βιώσιμο και το οποίο θα αντιτίθεται στη σπατάλη των τροφίμων. Βεβαίως οι πρώτοι που θα πρέπει να δείξουν το καλό παράδειγμα θα πρέπει να είναι τα ευρωπαϊκά όργανα ξεκινώντας από τούτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προωθήσουμε μια πραγματική εκστρατεία ευαισθητοποίησης ε, με μπροστάριδες πάντα τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Μια ε, καμπάνια, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που θα ε, μας οδηγήσει σε ένα πιο αηφόρο και μετριοπαθές μοντέλο κατανάλωσης. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίξαμε το ρόλο μας. Τώρα ευελπιστούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζοντα το δικό της θα οδηγήσει ε, σε μια συγκεκριμένη σειρά μέτρων. Ε, ε, πρώτα το 2014 να οριστεί Ευρωπαϊκό έτος κατά της πατάλης των τροφίμων. Αυτό θα καταδείξει άμεσα την δέσμευση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να δείξουμε σε όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είμαστε οι πρώτοι που ότι θα πρέπει να αλλάξει το κοινωνικό μοντέλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με το Catch the Eye πρέπει να ολοκληρώσουμε σε 15 λεπτά ούτως ώστε και ο Επίτροπος να απαντήσει εγκαίρως και να μην κρυφτεί η φωνή του πίσω από τον θόρυβο των συναδέλφων που θα έρθουν πριν τις 12 για, να, για τις ψηφοφορίες. Ο κύριος Λαβία καταρχάς. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε περαιτέρω αύξηση της πατάλης των τροφίμων. Θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και μέσα από μια αλλαγή πολιτισμική. Ε, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει σπατάλη. Αυτή η σπατάλη που αυξήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια κατά 50% με μεγάλες κοινωνικές, ε, ε, δεοντολογικές, ηθικές, αλλά και περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. 70 περίπου εκατομμύρια στην Ευρώπη ζουν κάτω από το όριο της ένδυας και είναι απαράδεκτο την ίδια στιγμή να υπάρχουν εκατοντάδες τόνοι αχρησιμοποίητων καλών τροφίμων που ρίχνονται στις χωματερές ή στα σκουπίδια θα πρέπει ε, να καταλάβουμε ότι η σπατάλη των τροφίμων σημαίνει και οικονομικό και κοινωνικό υψηλό κόστος. Ε, θα πρέπει να, δοθούν, να, υπάρξουν νέα μέτρα και όσον αφορά την ημερομηνία ε, λήξης των προϊόντων και όσον αφορά άλλα συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τικάου. να σας υπενθυμίσω ότι όποιος παίρνει το λόγο στο Catch the Eye για ένα συγκεκριμένο θέμα δεν θα πρέπει να πάρει το λόγο για το επόμενο θέμα. Δεν θα το εφαρμόσω βέβαια αυστηρά αυτό, αλλά θέλω να σας καλέσω όλους να είστε εξαιρετικά σύντομοι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα ότι στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 179 τόνους ανακάτοικο ε, τρόφιμα τα οποία σπαταλιώνται και πετιώνται. Ταυτοχρόνως πάρα πολλοί άνθρωποι διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. 16 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από την ενίσχυση και την βοήθεια των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε μια υγιεινή, επαρκή διατροφή. Το πρόβλημα της πατάλης των τροφίμων πρέπει να το προσεγγίσουμε λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υιοθετήσει πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ε, μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό, όπως δίνει ε, στο θέμα της ενεργειακής επάρκειας. Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα τη πατάλη των τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι ασχολείται με το θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πόσο μάλλον εφόσον υπάρχουν πραγματικά καταστροφικέ προγνώσει όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των τροφίμων και σε σχέση με τις ε, δημογραφικές εξελίξεις. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται επίσης ε, με τα όσα συζητούμε εδώ, με άλλους τομείς δηλαδή, με το εμπόριο, με το λιανικό εμπόριο τροφίμων και εδώ υπάρχει εκτεταμένη σπατάλη τροφίμων γιατί τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορούν να πωλήσουν. Όπως είπαμε, η σπατάλη των τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν θα πρέπει να την παραγνωρίζουμε όταν συζητούμε για την, για την υπερεκμετάλλευση των ε, γεωργικών εκτάσεων. Κύριος Νικολάσικ. Ε, ναι, Ε, σπαταλώνται πάρα πολλά κιλά ε, τροφίμων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός και θα πρέπει να συμπεριληφθεί μεταξύ των προτεραιοτήτων μας. Ε, τα πιο φτωχά τμήματα του πληθυσμού πλήττονται από αυτό το φαινόμενο, εξίσου όπως και το περιβάλλον. Και αυτό επιφέρει σημαντικές απώλειες για τις επιχειρήσεις αλλά και για ολόκληρη την οικονομία. Ένας εξορθολογισμός της ε, αλυσίδας, ε, διανομής, αποθήκευσης κλπ ε, θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση γιατί πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες τροφίμων χάνονται. Γι' αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε μια σύνθετη ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτή την κατεύθυνση. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε που ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτό. Κυρία Μακίνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετική ιδέα πραγματικά να προσέξουμε ιδιαίτερο στο ζήτημα αυτό και προτείνουμε ε, το έτος 2004 να είναι ένα έτος που ε, το 2014 να είναι ένα έτος το οποίο ε, θα είναι αφιερωμένο στο θέμα αυτό. Είναι και έτος εκλογών άλλωστε. Δεν γίνεται λόγος μόνο για τα τρόφιμα που πετάει ο καθένας σπίτι του, αλλά και αυτό εδώ το θεσμικό όργανο, τα νοσοκομεία, οι δημόσιοι φορείς σπαταλούν πάρα πολλά τρόφιμα. Και όλα αυτά που είπαμε ταιριάζουν με αυτά που είπαμε προηγουμένως για την αλυσίδα ε, προμήθειας ε, τροφίμων. Εάν μειώσουμε τα τρόφιμα που πετιόνται θα έχουμε ε, μια πιο βιώσιμη κατάσταση. Ευχαριστώ η κυρία Πρέντεργκαστ. Ευχαριστώ πολύ. 7 δις έφτασε ο πληθυσμός της γης ε, και το 2015 μάλλον 50 ε, θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια. Επομένως η επισητιστική ασφάλεια είναι ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα εστιάζοντας την παραγωγή περισσότερης τροφής για τον άνθρωπο θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε τους τρόπους μείωσης της σπατάλης των ε, τροφίμων. Η σπατάλη γίνεται σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής, από την παραγωγή δηλαδή μέχρι την τελική κατανάλωση. Αλλά βεβαίως ε, οι διαφορές ε, είναι σημαντικές ανάλογα με τη χώρα. Στις προηγμένες χώρες η σπατάλη γίνεται στο τέλος της αλυσίδας, ενώ αντίθετα στις αναπτυσσόμενες στην αρχή της αλυσίδας. Στην ε, Ιρλανδία ε, έχουν ε, ληφθεί συγκεκριμένε δράσεις όπως ας πούμε το Stop Waste Food ή μια αλυσίδα αλληλεγγύης που βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νιπουλέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εξοικονόμηση τροφίμων σημαίνει εξοικονόμηση εργασίας, εξοικονόμηση ε, οικονομικών πόρων και άλλων πόρων. Συζητήσαμε πολύ τελευταία το θέμα της ε, γεωργίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται πολύ από γεές ε, οι οποίες βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Χρησιμοποιεί κάθε χρόνο 640 εκατομμύρια εκταρίων γεών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται ε, στην ουσία 10 φορές ε, για, μια ε, επιφάνεια 10 φορές μεγαλύτερη από τη Γερμανία. Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας γιατί πλέον είναι δυσέβρετοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ο κύριος Κουμουτσάκος δεν είναι εδώ κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γκαρόνα γιατί ε, με πολύ σωστό τρόπο παρουσίασε το ζήτημα αυτό κάτω από το πρίσμα του κοινωνικού σκανδάλου αλλά και κάτω από ε, άλλες κοινωνικές και οικονομικές ε, πλευρές που σχετίζονται με της τροφίμων Θα ήθελα λοιπόν να στραφώ προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ταγιάννη, για να το ρωτήσω το εξή. τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα κατά της σπατάλης, πώς είναι δυνατόν ε, να εξευρεθούν κεφάλαια και κονδύλια τα οποία θα αφιερωθούν στον σκοπό αυτό πρέπει ε, να ε, ε μπορέσουμε ε, είτε μέσα από το Κοινωνικό Ταμείο είτε μέσα από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να χρησιμοποιήσουμε και την αλυσίδα γεωργικής παραγωγής έτσι ώστε όλα τα συμβαλόμενα μέρη διακόπτεται ο κύριος Μάουρη, η κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε εποχές ε, κρίσης και περικοπών δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι 50% των ε, τροφίμων τελικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Συγητή που αφιέρωσε την προσοχή του σε αυτό το θέμα. Και η νομοθετική εξουσία χρεώνεται αυτή την αποτυχία. Η παραγωγή δεν ε, έχουν στη διάθεσή τους από την άλλη αρκετές ε, πληροφορίες. Πολύ ε, πολλές φορές αναγράφονται πολύ σύντομες ημερομηνίε λήξης των προϊόντων και αυτό θα πρέπει να αλλάξει ε, λυπούμε λοιπόν, που παραλείπονται να αναφερθούν οι τράπεζε τροφίμων στην έκθεση. Πρόκειται για μη κυβερνητικού οργανισμούς που ασχολούνται με τη διανομή τροφίμων στα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για την ε, βοήθεια σε τρόμα και νομίζω ότι αυτή η τράπεζα θα μπορούσε να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πετούμε ουσιαστικά το 1 τέταρτο αυτών που ψωνίζομαι. Ε, οικονομικά και ηθικώς είναι παράδεκτο. Ο καθένας μας μπορεί κάτι να κάνει γι' αυτό, στην κουζίνα του, στο σπίτι του, όταν κάνει τα ψώνια του. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε καλύτερα τον κόσμο και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκύψει πάνω στο θέμα αυτό. Μιλούμε για την διατροφική επάρκεια μόνο και όχι μόνο την ποιότητα πάρα πολλοί κρίκοι της διατροφικής αλυσίδας θα γίνουν πολύ πιο ισχυροί. Τα τρόφιμα θα διαρκούν και περισσότερο. Θα ήθελα και ο, ο, κλάδος των τροφίμων να αναλάβει τις δικές του ευθύνες που του αναλογούν για τους εκατομμύρια Ευρωπαίους. Οφείλουμε να επιστρέψουμε στην αγροτική κουλτούρα, να είμαστε πιο ευαίσθητοι έναντι αυτών που καταναλώνουμε. Θα πρέπει να αξιοποιούμε τα υπολείμματα των τροφίμων και να μην τα πετάμε με το παραμικρό. Ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye. Θα δώσουμε το λόγο στον ε, Επίτροπο κύριο Ταγιάννη. Ως πρώην συνάδελφος κύριε Ταγιάννη, σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος και εσείς, έτσι ώστε ε, να, μην, να προλάβουμε να μην μπουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και τελικά δεν ακούγεστε στην αίθουσά σας. Θα ήθελα να μην ξεπεράσετε τα 5 ή 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Βλέπω ότι και ο κύριος Βόμποντα είναι ε, στη θέση του, γι' αυτό θα ήθελα να του εκφράσω τις ε, καλύτερες ευχές μου για τη νέα του θέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Καρόνα, τον εισηγητή, καθώς επίσης και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Εσωτερικής Αγοράς για το θέμα αυτό. Ο ε, Επίτροπος που είναι υπεύθυνο για τη γεωργική πολιτική και ο οποίος δεν είναι εδώ γιατί βρίσκεται στο Δουβλίνο, έτσι ώστε να παρουσιάσει την κοινή γεωργική ε, ε, πολιτική εις την Ιρλανδία. Και τον εκπροσωπώ εγώ. Το θέμα τη ε, επιστηστικής Αλυσίδα και διατροφική επάρκεια είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά και εκεί παίζει σημαντικό ρόλο το θέμα τη σπατάλης. Κατά αυτή την έννοια θα ήθελα να αναφερθώ στη διάσκεψη που έλαβε χώρα την 28 Οκτωβρίου 2010 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω, τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει πολλέ προτάσει. Και εκπονεί πληθώρα άλλων έτσι ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό το πρόβλημα της πατάλης των τροφίμων και αυτό μάλιστα σε διάφορα επίπεδα. Ε, ήδη αναφέρθηκα στην ε, διαμόρφωση, στη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ που αφορά βεβαίως και την παραγωγή αλλά και την μεταποίηση. Τα μέτρα σε ισχύ τα οποία θα κάνουν πιο αηφόρο τον τομέα όλα αυτά δηλαδή τα προγράμματα τα οποία βοηθούν κατά αυτή την έννοια θα διατηρηθούν. Επίσης για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις άλλες προτάσεις που υποβάλλει η έκθεση ε, όπως ας πούμε ε, υποπρογράμματα θεματικά στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου βάσει των οποίων θα δημιουργηθούν πολύ βραχίες αλυσίδες διατροφικής επάρκειας έτσι ώστε να μειωθεί η σπατάλη. Βεβαίως η καινοτομία όσον αφορά και την παραγωγή αλλά και την αηφόρο ανάπτυξη στη γεωργία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό θέλουμε αηφόρο γεωργία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους. Το φόρουμ υψηλού επίπεδου όσον αφορά την επισητιστική αλυσίδα ε, του, για το οποίο συζητήσαμε ήδη σήμερα το πρωί εργάζεται ε, και για τα θέματα της βέλτιστης πολιτικής όσον αφορά τις συσκευασίες και όσον αφορά τις ημερομηνίες ανάλωσης των προϊόντων. Ε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ε, και σε συνεργασία και με την Στρογγυλή Τράπεζα για την αηφόρο ανάπτυξη συνεργάζεται λέω με όλους αυτούς τους φορείς έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αποτελέσματα. Τον ε, Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξεπώνησε ανακοίνωση όσον αφορά την γεωργική ανάπτυξη και την επιστημική αλυσίδα μέχρι το 2050. Είναι γεγονός ότι τα τρόφιμα αποτελούν έναν από τους κυριότερους φορείς που μπορούν να μας βοηθήσουν στην ε, καλύτερη χρήση των πόρων. Ε, ο δικός χάρτης που καθορίζει πολλούς φιλόδοξου στόχους όσον αφορά τη μείωση σπατάλης των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 ε, έχει στόχο να φτάσει σε μείωση της, της τάξης του 20% των ε, πρώτων υλών. Ε, και των πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ε, τροφίμων. Το 2003 θα υπάρξει ανακοίνωση για την αηφόρο διατροφή έτσι ώστε να προχωρήσει και να προωθήσουμε με συνεκτικό και ε, σωστό ορθό τρόπο αυτό το σημαντικό ζήτημα. Μεθοδολογία η οποία θα βασίζεται σε κριτήρια βιωσιμότητας μέχρι το 2014. Σε μία από τις ε, συστάσεις σας, ε, την υπαριθμό 35, ζητάτε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ορίσουν το 2013, λέει ο Επίτροπος, το, Ευρωπαϊκό έτος κατά της σπατάλης. Ο Επίτροπος Νταλή θα συζητήσει το ζήτημα αυτό με τον εισηγητή σας, γιατί όλοι συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η σπατάλη των τροφίμων στο σύνολο της διατροφικής αλυσίδας. Όμως το 2013 είναι πρόημο. Πρώτον γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει προτείνει ήδη για το 2013 να οριστεί σαν Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Επίσης γιατί χρειαζόμαστε περίπου δύο χρόνια έτσι ώστε να προετοιμάσουμε σωστά και από όλε τις πλευρές ένα Ευρωπαϊκό Έτος στις συζητήσεις γίνεται λόγος από ό,τι καταλαβαίνω ε, ε, λέει ο, ο κύριος Επίτροπος ε, μιλάτε για το 2014 και όχι για το 2013 αυτό ίσως να είναι πιο εφικτό αλλά βεβαίως θα πρέπει να μιλήσω με τους δύο συναρμόδιους επιτρόπους έτσι ώστε να δούμε εάν και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι δυνατόν αυτά ήθελα να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε κύριε Σιγητά κυρίες και κύριοι για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όσοι ζήτησαν το λόγο μετά την έναρξη του Catch the Eye δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο διότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν όλοι σύντομοι. Έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να απεφευχθεί τη δυσάρεστη εξέλιξη του να μην είμαστε σε θέση να ακούσουμε τον Επίτροπο από το θόρυβο των υπολείπων που μπαίνουν στην αίθουσα για να ψηφίσουν. Θα διακόψουμε τώρα τη συνεδρίαση για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες στις 12 το μεσημέρι ακριβώς.